ευρωπαϊκού κειμένου, διότι δίνουμε μια άλλη δυνατότητα ελέγχου των εξουσιών ε, των θεσμικών οργάνων. Ο κανονισμός για την πρωτοβουλία πολιτών που υιοθετήθηκε με την συνήθι νομοθετική διαδικασία έχει ως στόχο να παράσχει στους πολίτες μας τα ίδια δικαιώματα πολιτικής πρωτοβουλίας που έχουν ήδη το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα εκατομμύριο υπογραφές χρειάζονται, δηλαδή 2% των πολιτών μας, για να καλέσει την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε τομείς που τους αφορούν ευθέως. Τους επιτρέπει να ακουστούν και θα δημιουργήσει άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καλύπτοντας το κενό που υπάρχει μεταξύ τους, μεταξύ όλων ημών και της κοινή γνώμης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αγωνίστηκαν σκληρά για να προχωρήσει γρήγορα η έγκριση του κειμένου αυτού σε πρώτη ανάγνωση και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία τις διάφορες προεδρίες, ιδίω δε τις προεδρίες του Βελγίου και της Ουγγαρίας, την Επιτροπή, τα μέλη του Κοινοβουλίου, ιδίω τους προέδρους των Επιτροπών Συνταγματικών Υποθέσεων και Αναφορών, τον κύριο Κασίνη και την Ερμήνια Ματσόνη αν θέλετε, ελάτε εδώ μπροστά να είστε παρόντες κατά τη διαδικασία υπογραφής. Τους τέσσερις εισηγητές, κύριο Λαμασούρ, Ζήτα Γκομάη, Νταϊάννα Γόλης και Γκέρατ Χέφνερ. Ελπίζω να είστε παρόντες, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία μαζί. Αλλά και όλα τα άλλα μέλη και σκιώδεις εισηγητές που μπορεί να είναι περήφανοι για το έργο που έχει καταβληθεί για τους πολίτες μας. Το Συμβούλιο θα υπογράψει τώρα το σχέδιο αυτό. Πριν από αυτό, ωστόσο, να ζητήσω από τους προσκεκλημένους μας, τον Προεδρεύοντα, για το εξάμεινο αυτό κύριο Μαρτώνη Υπουργό, να πει δύο λόγια. Κυρίες και κύριοι, Στη συγκινητική αυτή στιγμή θα ήθελα να θυμίσω τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Συνθήκης όταν συνέλευσης, όταν μιλούσαμε για το δημοκρατικό έλλειμμα της ε, διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και συζητούσαμε πώς θα μπορούσε να μειωθεί. Είχαμε έναν κοινό στόχο να ενισχυθεί η δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης. Ε, και γι' αυτό θελήσαμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Γι' αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών έχει συμπεριληφθεί στη συνθήκη και τώρα έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν απευθείας στην Κομισιόν για να ζητήσουν την υποβολή νομοσχεδίου. Πιστεύω ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό βήμα στο δρόμο προς την αύξηση της δημοκρατικότητας της Ένωσης και είναι το πρώτο στοιχείο άμεσης δημοκρατίας γιατί καθορίζει έναν διάλογο μη μεσολαβημένο μεταξύ θεσμικών οργάνων και πολιτών. Ενθαρρύνει τη διαμεθοριακή συνεργασία. Επίσης, ενθαρρύνει το αίσθημα ιδιοκτησίας της Ένωσης από τους πολίτες. Η Ένωση δεν βλέπει, δεν θεωρείται πια σαν οι άλλοι αλλά σαν εμείς και μάλιστα όλοι εμείς. Το σύνθημά μας ισχυρή Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο εξαρτάται από όλους μας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και για να εφαρμοστεί σωστά η συνθήκη χρειάζεται χρειάζονται σαφείς και φιλικοί προς το χρήστη κανόνες. Πράγμα το οποίο πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας με όλα, όλων των θεσμικών οργάνων, δηλαδή Συμβουλίου, Κοινοβουλίου κυρίως και Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Σεύκοβιτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης τις ευχαριστίες μου στην Ισπανική και Βελγική Προεδρίες και ιδιαιτέρως, ιδιαιτάτως ευχαριστίες και συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλους όσους συμμετέσχουν σε αυτήν τη σημαντικότατη δουλειά, τον πρόεδρο, τον, τους πρόεδρους των Επιτροπών και τους εισηγητές και εισηγήτριες Λαμασούρ, Ζήτα Γκούρμαϊ, Ναναβόλης, Χέφνερ και όλα τους άλλους βουλευτάς που συμμετέσχουν σε αυτή την πολύτιμη εργασία που δείχνει πόσο σημαντική και αποτελεσματική μπορεί να είναι η συνεργασία και η κατανόηση όχι μόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και μεταξύ των διαφόρων πολιτικών οικογενειών ή ομάδων. Και δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ελπίδα μου η συνεργασία και η κατανόηση αυτή να αποτελέσουν πρότυπο για το μέλλον και για τα θεσμικά όργανα και για τις πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Τώρα θα γίνει η διαδικασία υπογραφής του νομοθετικού κειμένου. La Presidente. Η Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η